Good evening everyone. Hello. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε στην έκτακτη σημερινή μας συνεδρίαση. Υποθέτω ότι συμφωνείτε με το σχέδιο μεσής διάταξης. Ε, δεν βλέπω να διαφωνεί κανείς. Έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες και ως ήθιστε μεταδίδεται απευθείας από το διαδίκτυο συνεδρίασή μας. έχετε λάβει και τις συστάσεις των συντονιστών στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και αν δεν διαφωνείτε θεωρούνται εγκεκριμένες. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω εξ ονόματός σας τώρα τον Επίτροπο, τον κύριο Άρια Σκανιέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κύριε Επίτροπε. Πρόκειται ε, για μια συνεδρίαση στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε ε, τις προτεραιότητές τους για το 2018 και το χειμερινό πακέτο ε, που έχουμε και εμείς στη μέση διάταξή μας και να μάθουμε και τις εξελίξεις και τα τεκτενόμενα για, για τις προσδοκίες σας ενδεχομένως για την επόμενη συνεδρίαση COP για το κλίμα. και τις τρέχουσες εργασίες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε και θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε καλέσατε να τα συζητήσουμε σήμερα όσον αφορά τις προτεραιότητες για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική στιγμή όσον αφορά την τήρηση των όσων υποσχεθήκαμε σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων και την υλοποίηση του πλαισίου για το κλίμα και την του 2030. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ την Επιτροπή και κυρίως τον Ιαν Τάγκαν τον εισηγητή αλλά και τους χειώδες για την πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά την πρόταση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS. Ήταν η διαδικασία ε, δύσκολη, εντατική στο Κοινοβούλιο και όλοι έπρεπε να συμβαστούν, αλλά πιστεύω ότι καταφέραμε να πετύχουμε μια δίκαιη λύση για την εντολή του Φεβρουάριο και έτσι νομίζω ότι δόθηκε μια όθηση που όπως χρειαζόταν για να εξασφαλιστεί ε, ε, η σύμβουλη γνώμη του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης χαίρομαι που ο τριμερής διολόγος πρόκειται να ξεκινήσει και επίσης πρόκειται να πετύχουμε, ελπίζω, να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις για το ETS το συντομότερο. Έχουμε τώρα την κοινή δήλωση για τις προτεραιότητες, οπότε είπαμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί ε, να ισχύει το για τις ε, πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπάρχει κάποια σαφήνεια όσον αφορά την εφαρμογή των ε, συμφωνιών για την Διεθνή Συμφωνία αυτό που ονομάζουμε Κόρσια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε σύντομα αυτή τη διαδικασία και ελπίζω ότι το Συμβούλιο αλλά και το Συμβούλιο πρόκειται μέχρι το τέλος του 2017 να έχουν συμφωνήσει πολύ πριν φτάσουμε στον ε, κύκλο ε, στην συμπλήρωση του κύκλου τέλο πάντων ε, συμμόρφωση το 2018. Επίσης να έχουμε τις προτεραιότητες 2017 στα πλαίσια αυτά. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα για τα άλλα στοιχεία του πλαισίου για κλίμα και ενέργεια όσον αφορά το πακέτο καθαρή ενέργεια όλους τους Ευρωπαίους και επίσης έχουμε τώρα το LLCF ε, όσον αφορά την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές Χερμπράντι και Λίνς για την πρόοδο που έχουμε πετύχει όσον αφορά την ε, ε, κατανομή της ευθύνης προσπάθειας και του LLCF και γενικά για το πόσο στήριξε την Επιτροπή. Οπότε ελπίζουμε ότι θα αρχίσουμε την υλοποίηση των υποσχέσεών μας του Παρίου ε, το καλοκαίρι και θα έχουμε τελειώσει τη διαδρομή τέλος του έτους και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα πλαίσια των μεταφορών και τι θα γίνει με, αυτό, με αυτή την δέσμη Clean Energy for All Europeans με αυτή την σημαντική δέσμη μέτρων θα προσπαθήσουμε να μείνουμε πρωτοπόροι όσον αφορά αυτή την ε, μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και θα υλοποιήσουμε τη Συμφωνία των ε, Παρισίων και θα καλύψουμε από αποτελεσματική χρήση ενέργειας, ανανεώσιμη ενέργεια και τον σχεδιασμό, προγραμματισμό ενεργικής αγοράς αλλά και τους κανόνες διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση. Έτσι, να έχουμε ένα πλαίσιο ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να εξοπλίσουν τις δυνατότητές τους όσον αφορά τα ανανεώσιμα και να φτάσουμε στο 27% ε, όσον αφορά τη χρήση των ανανεώσιμων στην ε, Ένωση ε, μέχρι το 2030 με καλή σχέση κόστους αποτελέσματος οπότε έτσι θα είμαστε πρωτοπόροι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους καταναλωτές και θα πετύχουμε να έχουμε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Οπότε θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει με τους στόχους του 2030 για να νεώσουμε και ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Επίσης για να έχουμε μια στιβαρή διακυβέρνηση θα πρέπει να συμβαστούμε, να ε, ε, υλοποιήσουμε τα όσα επιτάσσει η συνθήκη των Παρισίων. Οπότε θα πρέπει έτσι να αρχίσουμε σύντομα τις σχετικές συζητήσεις και το Κοινοβούλιο θα πρέπει το συντομότερο να διαδραματίσει το ρόλο του για αυτό το πλαίσιο, ούτω ώστε να έχουμε ε, την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων προγραμμάτων για το κλίμα και την ενέργεια σε επίπεδο εθνικό. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες προσπάθειες φιλόδοξες αλλά και συγκεκριμένες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, η πρωτοβουλία για το πακέτο καθαρής ενέργειας ε, είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτό και θα προχωρήσουν αυτά χέρι-χέρι κατά τη διαδικασία συναπόφασης. Εσείς θα πρέπει να βοηθήσετε. Και τώρα, δύο λόγια για τις οδικές μεταφορές. Είναι το 25% των εκπομπών μας, άρα χρειάζεται μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και αυτό αποτελεί και αντικείμενο της Συμφωνίας των Παρισίων. Τέτοια ε, συμφωνία, τέτοια στρατηγική χρειάζεται. Γι' αυτό και πέρσι τον Ιούλιο ξεκινήσαμε με αυτή τη δέσμη μέτρων. Καθαρή συνεργασία για του Ευρωπαίου. Οπότε η αναβάπτιση τη σχετική οδηγία για τα ανανεώσιμα δίνει κίνητρα για ανανεώσιμα καύσιμα. Χρειάζεται επομένω αυτή η εντολή ενσωμάτωση. Αυτό προτείνουμε ούτω ώστε να έχουμε όλο ένα περισσότερη συμμετοχή καυσίμων ανανεώσιμων αλλά και βιοκαύσιμα. Έχουμε προτείνει κάποιες ε, τροποποίησεις στην οδηγία για η ηλεκτροκινητικότητα και επίσης ε, έχουμε μια στρατηγική για ΕΦΗ e συστήματα μεταφορών που διακρίνονται από συνεργασία CITS και αυτό θα βοηθήσει την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, οικολογική οδήγηση και μείωση του δεξιδίου. Επίσης ετοιμάζω μονοθεσία και αυτό θα γίνει αργό το 2017, νέους στόχους για εκπομπές διοξιδίου και επίσης να έχουμε κάποια οχήματα χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών. Οπότε έτσι θα βοηθήσουμε στο να υπάρχει αυτή η μετάβαση για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Οπότε η μελέτη επιπτώσεων θα μας δείξει κόστη, κέρδη διαφορετικών επιλογών, να δούμε τι γίνεται με το χρονισμό, το timing και τι κίνητρα θα υπάρχουν για αυτά τα ε, οχήματα χαμηλών εκπομπών. Όλοι αυτοί οι στόχοι με το 2020 θα βασίζονται στη διαδικασία των δοκιμών του παγκόσμιου χαρακτήρα για οχήματα ελαφρά. Και έτσι θα έχουμε πιο ρεαλιστική κατανάλωση και επίση εκπομπές. Επίσης του χρόνου πρόκειται να προτείνουμε κάποια πρότυπα για τις εκπομπές. Αναλυτική εργασία γίνεται τώρα για όλα αυτά τα οχήματα. Πρώτα όλα όμω χρειάζεται κάποιο είδου πιστοποίηση για διοξείδιο του άνθρακος και θα πρέπει να γίνει έλεγχη, εποπτεία όσον αφορά τα βαρέα <clears throat> οχήματα και όλα αυτά θα εγκριθούν πριν το θέρος. Εάν επομένως βοηθήσουμε τη δράση των κρατών μελών, αυτό θα είναι βασικός πυλώνας για την στρατηγική προσαρμογή που αποφασίζεται το 2013 και έτσι θα υλοποιήσουμε τη σχετική στρατηγική και θα προτείνουμε μια σχετική έκθεση για Κοινοβούλιο και Συμβούλιο μέσα του 2018. Με αυτή την έκθεση επίσης θα επισυνάψουμε και μια στρατηγική αναθεωρημένη, στρατηγική προσαρμογής που να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, τις συνέπειες της Συμφωνία των Παρισίων, ούτω ώστε η δράση μας να προσαρμοστεί με τα όσα γίνονται εντός και εκτός των συνόρων και οι διαβουλεύσεις το 2017 θα λάβουν χώρα δύο εργαστήρια αρχά Απριλίου και Σεπτεμβρίου και κάποια διαβούλευση ε, Ιντερνετική Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο. Τώρα όσον αφορά την αυτιλία αφού εγκρίθηκε το Παγκόσμιο Σύστημα Συλλογή Δεδομένων όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων από τα πλοία από τον ΆΕΜΟ Οκτώβριο του 2016, ετοιμάζουμε την αναθεώρηση, την αξιολόγηση του κανονισμού για την παρακολούθηση τις εκθέσεις, την παλήθευση των εκπομπών από μεταφορές που λέγεται κανονισμός MRV. Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σύστημα του IMO, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, αλλά επίσης και την επαλήθευση των δεδομένων που είναι βασικά στοιχεία του κανονισμού μας. Εάν χρειαστεί, πρόκειται να κατεβάσουμε αυτή πρόταση για να τροποποιηθεί αυτός ο κανονισμός MRV, όσο χρειάζεται του πρώτου ημίση του 18. Αυτό θα αλλάζει χώρα εκ παραλίλου με συζητήσει τον ΑΕΜΟ για κάποια στρατηγική μείωση των εκπομπών για την διεθνή ναυτιλία που πρόκειται να εγκριθεί την άνοιξη του 18. Ε, επίσης θα έχουμε κάποιου στόχου ε, φιλόδοξου για μείωση των εκπομπών και να πάμε πιο κάτω από το στόχο των 2 βαθμών Κελσίου. Όλα αυτά θα συζητήσουμε και για να δούμε τώρα τι γίνεται διεθνώ όσον αφορά το κλίμα του χρόνου. Θα είναι μια χρονιά πολύ κρίσιμη για τι διαπραγματεύσει παγκοσμίω. Έχουμε όλου αυτού του ενδελεχεί κανόνε Συμφωνία των Παρισίων που τώρα είναι διαπραγμάτευση και πρόκειται να εγκριθούν στο COP24 του 18. Επίση, τότε στο COP24 του 18 πρόκειται να έχουμε τον διάλογο διευκόλυνση όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγηση που θα ευθυγραμμιστεί με το όραμα και τους μακρόπνους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων που θα είναι η επόμενη σημαντική καμπή και παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις θα εντείνουμε προσπάθειες για να έχουμε ε, υλοποίηση των εθνικών στόχων αλλά και των στόχων των εταίρων μας επίσης να εντείνουμε τη διπλωματία μας και η οικονομική υποστήριξη στις πιο φτωχές χώρες και αυτό θα γίνει με διάλογο, με ζήμωση κυρίως στο G20 που ευθύνονται 180% των κομπών και είναι πολύ θετικό το ότι στο Συμβούλιο των Υποθέσεων τη Έκτη Τρίτο, επαναναλήφθηκε το ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμπεράσματα αυτά και θα πρέπει οι πιο σημαντικέ οικονομίε να κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα των Παρισίων και πρόκειται για μια συγκυρία διεθνή πολύ προβληματική, αλλά και είναι και πρόκληση και να συνεχίσουμε να δείχνουμε, να βάλουμε δράση, ότι είμαστε αποφασιστικοί να υλοποιήσουμε το ότι συμφωνήσαμε, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη βιομηχανία, με τι πόλει, με όλου εμπλεκόμενου στα πλαίσια του θεματολόγιου τη δράση για το κλίμα και να ενθαρρύνουμε επενδύσεις, απασχόληση και να έχουμε απτά για τον κόσμο. Όπως βλέπετε είναι πλήρες το θεματολογιό μας για το κλίμα και την ενέργεια και γεμάτο πρωτοβουλίες του χρόνου και θα περιμένω πώς και πώς το πώς θα συνεργαστούμε φέτος και πώς θα αναβαθμίσουμε το διάλογο και θα κάνουμε περαιτέρω διαδήματα για την υλοποίηση των όσων υποσχεθήκαμε στο Παρίσι. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Όσοι ήθιστε, οι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο να σχολιάσουν, να κάνουν ερωτήσεις. Αρχίζουμε το πρώτο γύρο συντονιστές. Θα ομαδοποιήσουμε τις απαντήσεις. Ο κύριος Λίζε, εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας και την προσήλωσή σε στην εργασία αυτή. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο σύστημα εμπορία εκπομπών ρήπων, ETS. Λάβαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από το Συμβούλιο και νομίζω ουσιαστικά πήγαμε στην ίδια κατεύθυνση ε, το Κοινοβούλιο. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρούμε πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα carbon leakage. Και χαιρετίζουμε την πρόταση του Συμβουλίου που θέλει να δίνει δωρεάν άδειε ε, στα εργοστάσια που βρίσκονται στην τελευταία λέξη της ε, τεχνολογίας και προτείνει 5% το Κοινοβούλιο και 2% το Συμβούλιο. Στην εκθεσία Αντάνκαν έχουμε αποφασίσει ε, και για τις αερομεταφορές και θέλουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Και με λίγη καλή θέληση νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε τελικά για αυτά που θέλει ε, φέρω μεταφορές στο Κοινοβούλιο για να αποφύγουμε και το carbon leakage στις ενεργοβόρες βιομηχανίες θα παρακαλούσα να το κοιτάξετε αυτό με τις υπηρεσίες σας. Χρειάζεται κάποιες προσαρμογές, γιατί θα έχει το πλεονέκτημα να μην ξαναπέσουμε στο παλιό παιχνίδι των επιχειρημάτων ε, των Υπουργών Μεταφορών απέναντι στους Υπουργούς ε, Περιβάλλοντος. Τώρα θα μπορούσαν να μας υποστηρίξουν ακόμα και οι Υπουργοί Οικονομικών στην εξισορροπημένη προσέγγιση. Στη συνέχεια, ε, πολύ σύντομα, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζητούν ε, μεγαλύτερη φιλοδοξία για την ακύρωση κάποιων ε, πιστοποιητικών. Τώρα όμως λυπάμαι ε, γιατί βλέπω ότι στον επιμερισμό των βαρών υπάρχει μία προσπάθεια λιγότερο φιλόδοξη. Έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο είναι λιγότερο φιλόδοξο από το ETS και υπάρχουν πολλοί αποχρόντες λόγοι για να μην αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίζε. Η κυρία Ντάλη, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ που βρίσκεστε μαζί μας εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Για τους σοσιαλδημοκράτες ε, είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε σε πράξεις, ε, να μην μιλάμε μόνο, κυρίως όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό ισχύει και για το ETS. Βλέπουμε πολύ θετικά ότι το Συμβούλιο έδειξε και αυτό περισσότερες φιλοδοξίες ε, όσον αφορά τον ορισμό των στόχων, αλλά θέλω να κοιτάμε προς το μέλλον, να εστιαστούμε στην καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους και τη σχετική δέσμη μέτρων, στην οποία αναφερθήκατε, πιο συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν μιλάμε για στόχο τουλάχιστον 27% ως στόχο προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιλάμε για στόχο πανευρωπαϊκό. Πείτε μου πώς ε, ε, σκοπεύει η Κομισιόν να ε, εξασφαλίσει την εκπλήρωση του στόχου χωρίς να υπάρχουν εθνικά δεσμευτικοί στόχοι. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσετε την εξή ανησυχία ότι μπορεί να δράσει αποτρεπτικά η αποδυνάμωση του πλαισίου για τις ανένομες πηγές ενέργειας για τους επενδυτές επειδή θα είναι επίσης και δυσκολότερο για τα κράτη-μέλη να τα υποστηρίξουν. Ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να τους δοθεί η υποστήριξη που απαιτείται. Ένα άλλο θέμα, η Ιρλανδία. Πρόσφατα συμμετείχα σε μια διάσκεψη για την Ιρλανδία και το ρόλο της στην Ενεργειακή Ένωση και ειδικότερα σε αυτή τη δεσμή μέτρων διότι κομισιών αναφέρεται σε νησιά, συγγνώμη, όχι Ιρλανδία, σε νησιά. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν να επιτύχει αποτελέσματα, δηλαδή τα νησιά ειδικότερα τα απομακρυσμένα να πάψουν να είναι απομονωμένα ε, και να πάψουν να εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Και τέλος, αναφερθήκατε στον τομέα των μεταφορών. Πρόσφατα έγιναν συναντήσεις και στο Βερολίνο, όπου εσείς συμμετείχατε και αναφερθήκατε και στη στρατηγική της Κομισιόν για κινητικότητα χαμηλίων εκπομπών. Η χρονική στιγμή αυτή είναι ενδιαφέρουσα γιατί οι λομπίστες των βιομηχανιών επίσης πιέζουν για τα δικά τους συμφέροντα και όπου η δράση βέβαια στα κράτη-μέλη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ε, για το που βρίσκονται τα κράτη-μέλη, τα κυριότερα όσον αφορά την απαλλαγή ε, του τομέα των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, ε, ειδικότερα η Γερμανία αφού ήσασταν στο Βερολίνο. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη, η κυρία Γκέρλινγκ, εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ. Και είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Η έκθεση αυτή από τότε που εκδόθηκε με απασχόλησε. Έψαξα να βρω για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη των βιοκαυσίμων στο σύστημα και εγώ δυσκολεύομαι να βρω ανθρώπους που να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να παράγουν βιοκαύσιμα στο αναμενόμενο επίπεδο. Να σας ρωτήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα, έχουμε έναν επαρκή ορισμό των προηγουμένων βιοκαυσίμων. Θεωρείτε ότι ο σημερινός ορισμός είναι επαρκής. Θεωρείτε ότι κάνει αρκετά η Κομισιόν για να ενθάρρει την ανάπτυξή τους. Ή μήπω έφτιαξε απλά ένα κανονισμό. Κάνουμε δηλαδή ό,τι χρειάζεται ώστε να εφαρμοστούν, να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Και δεύτερον, μια ερώτηση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών για την αεροπλοεία. Η Επιτροπή έχει ασχοληθεί με αυτό, έχει κάνει πολλές επισκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα και διαρκώς ζητάμε πρόσβαση μεγαλύτερη στις ε, πληροφορίες, μεγαλύτερη διαφάνεια. Η DG Κλίμα μας διαβεβαίωσε ότι σίγουρα στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, ETS για την αεροπλοεία θα μπορέσουμε να βασιστούμε στην υποστήριξη της Γενικής Διευθύνσης για το κλίμα που θα μας κοινοποιήσουν τις διαδικασίες τους διότι αν αυτό δεν γίνει δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, στις προσπάθειες που κάνουμε για το ETS για την αεροπλοεία πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι πρόοδοι και με το σημερινό καθεστώς αδιαφάνειας αυτό είναι δύσκολο. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε αν έχει γίνει κάτι όσον αφορά αυτό το θέμα της διαφάνειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, ο κ. Μπραντικ, μέρος του Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Η πρώτη ερώτηση αφορά ε, την ε, συνειδητοποίηση και ε, την δημόσια και ιδιωτική ανάληψη της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ καλή στη δουλειά, ε, κάνει μελέτες αντικτύπου, χιλιάδες σελίδων δημοσιεύει, αν υπάρχει δεν υπάρχει το λεγόμενο carbon leakage, ε, ποιος τομέας πρέπει να παίρνει δωρεάν άδειε και πιστοποιητικά. Εκεί διαπρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά, η συνειδητοποίηση του κοινού, δημόσια και ιδιωτική για την επίγουσα κατάσταση και τον επίγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει τεράστιο πρόβλημα εκεί. Αν δω τι κάναμε ε, με το σύστημα εμπορία εκπομπών εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο, μπορούμε να πούμε ότι ήταν λίγο ε, χαμηλότερη η δική μας φιλοδοξία και υψηλότερη η φιλοδοξία του Συμβουλίου, αλλά στο τέλος έχουμε μια πολιτική διαδικασία που μάλλον προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες για να μην λάβουμε κάποια μέτρα παρά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πάρα πολύ σοβαρά και ε, ακόμα περισσότερα από ό,τι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε βάσει μελετών αντικτύπου και επιπτώσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμεί έχουμε εκλογέ μεθαύριο στην Ολλανδία. Και ο Ολλανδικός Οργανισμός Περιβάλλοντος ανέλησε όλα τα πολιτικά μανιφέστα όλων των κομμάτων. Και τρία κόμματα έχουν μανιφέστα που ε, αντέχουν στο Παρίσι. Χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες, όχι. Το μεγαλύτερο κόμμα, η συντηρητική φιλελεύθερη, το κόμμα της ελευθερίας του Χέρτ Φίλτερς, να μην τον αναφέρω καλύτερα καθόλου. Μόνο η πρασινη σοσιαλ φιλελεύθεροι και με ένα μικρό χριστιανικό κόμμα είχαν προγράμματα σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων. Εγώ δεν θέλω να τονίσω τη σημασία του δικού μου κόμματος ή των Πρασίνων. Αναπώ ότι δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση για την κλιματική αλλαγή ακόμα σε μια χώρα όπως είναι η Ολλανδία. Όλοι εστερνιζόμαστε εμεί στη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά τα ίδια μας τα πολιτικά μανιφέστα δεν συνάδουν. Αυτά λέει ο Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο αρμόδιος της Ολλανδίας. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα από τα τεχνικά εγχειρήματα για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κοινού ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά το διεθνές προσκήνιο. Ακούσαμε τις ε, ε διακηρύξεις του νέου διευθυντή του Περιβαλλοντικού Οργανισμού στις ΗΠΑ, ε, ο οποίος αμφιβάλλει κατά πόσο η ανθρώπινη δραστηριότητα και το διοξείδιο του άνθρακα ε, είναι οι αιτίε τη κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι ΙΠΑ, αλλά ξέρουμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα ε, στο διεθνέ προσκήνιο. Και ποιε είναι οι επαφέ που έχετε εσεί αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και μετά, δεύτερον, τι γίνεται με την Κίνα. Ε, επίκειται μια σύνοδο κορυφή με την Κίνα το Μάιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρο ότι το κλίμα θα συζητηθεί ω προτεραιότητα. Είστε έτοιμος να λάβετε το ρόλο που είχαν παίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία διετία ε, να συνεργαστείτε δηλαδή με κάποιο τρόπο με την Κίνα ώστε να προωθήσετε περαιτέρω τα θέματα του περιβάλλοντος παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκριμπράντη. Η κυρία Τόρες Μαρτίνες, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ δεν θα είμαι τόσο ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στον Επίτροπο. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει από 80 μέχρι 95% μέχρι το 50% ε, τα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα ε, με τα επίπεδα του 1990. Επίσης, 1,5 βαθμό Κελσίου μας δεσμεύει να μειώσουμε τους στόχους της Συμφωνία του Παρισίου. Πώς θέλετε να τα κάνετε αυτά κύριε Επίτροπε όταν κάνετε μεγάλους ε, αγωγούς ε, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις που πληρώνουν οι πολίτες και μάλιστα η ζωή τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 50 χρόνια. Εκεί έχουμε διαρροές μεθανίου στους αγωγούς φυσικού αερίου. Μειώνουμε έτσι ε, τις εκπομπές και το μεθάνιο μπορεί να ευθύνεται 86 φορές περισσότερο από το διοξίδιο του άνθρακα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θα πρέπει οι χώρες να βασίζονται σε μια ε, μετάβαση ε, από το ε, ανάνθρακα στο αέριο, το φυσικό αέριο. Εδώ πρόκειται για όργια επενδύσεων σε αγωγούς φυσικού αερίου και να με συμπαθάτε που το λέω έτσι, αλλά φέρετε να ενδιαφέρεστε εσείς πιο πολύ για τα συμφέροντα των ε, δικών σας ε, επιχειρήσεων και των φίλων σας ε, και για την, παραγωγή, την ίδια παραγωγή για ίδια κατανάλωση γνωρίζετε τι γίνεται στην Ισπανία, το κόμματό σας ε, έβαλε βέτο στο νόμο αυτό για την παραγωγή προς κατανάλωση. Είναι παράδοξο γιατί το άρθρο 21 της ε, οδηγίας για τις ανανεώσιμες από το χειμερινό πακέτο ακριβώς αυτό θέλει. Το άρθρο 21 λοιπόν ορίζει ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται ιδιαίτερα εγκαταστάσει παραγωγής ρεύματος για ίδια κατανάλωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν στα νοικοκυριά την αυτοκατανάλωση. Όπως γνωρίζετε, στο Ισπανικό κράτος δεν πληρείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα βασιλικό διάταγμα ε, το οποίο επιβαρύνει τα νοικοκυριά και ε, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπουν άλλες συμβατές. Τι θα κάνετε για να υποχρεώσετε το κόμμα σας, το Λαϊκό Κόμμα, να σεβαστεί ε, τα ευρωπαϊκά κεκτημένα και τις επιταγές. Ε, εγώ αμφιβάλλω να μου επιτρέψετε γιατί όπως εσείς όπως και οι δικοί σας συνάδελφοι φέρεστε εμπλεκόμενο σε πολλά σκάνδαλα επιχειρηματικά ε, και άλλα. Και για σας μιλάω για πράγματα που γνωρίζετε και για ξέπλυμα χρήματος, για τα Panama Papers, ακόμα και αν δεν με κοιτάζετε και εξακολουθείτε να στρέφετε το βλέμμα σας. Το πρόβλημα είστε εσείς και δικοί σας. Εδώ και καιρό δεν θα πρέπει να ήσασταν στα θεσμικά όργανα και να στρώνετε κόκκινα χαλιά στις μεγάλες εταιρείε ενώ καταστρέφετε εσεί τον πλανήτη μας και τα δικαιώματα του κόσμου. Ευχαριστούμε κυρία Τόρας Μαρτίνες. Ε, βγήκατε εκτός θέματος λίγο, αλλά δεχόμαστε. Κύριε το επόμενο ομιλητή εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εισαγωγική σα παρουσίαση. Να αναφερθώ σε ένα-δυο σημεία. Χαίρομαι που η ε, Πετρελίσσα έχει αντιληφθεί ότι το Συμβούλιο είναι πιο φιλόδοξο από το Κοινοβούλιο για το ETS. Το δελτίο τύπου σα ε, τα έλεγε κάπω διαφορετικά, αλλά καλό είναι που καταλήξατε σε άλλο συμπέρασμα στο μεταξύ. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη, ε, μπορείτε να απαντήσετε αργότερα, ε, αλλά... Νομίζω ότι καταλαβαίνω το ETS αρκετά καλά, ξέρετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θέλω με το ETS αυτή τη στιγμή, κάτι που θα ανησυχήσει και την Κομισιόν, είναι ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη συζητούν εθνικά μέτρα. Διότι το ETS δεν φέρνει αποτελέσματα. Αν δείτε την αναθεώρηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και συνδυάστε τις θέσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η μεταρρύθμιση δεν θα τιμολογήσει έτσι τον άνθρακα ώστε να δώσει κίνητρα για καινοτομία. Σε όλο και περισσότερες λοιπόν χώρες συζητούνται επιπλέον μέτρα. Οπότε η ερώτησή μου προς εσάς είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μετά από αυτό το γύρο των διαπραγματεύσεων ότι αυτό που φτιάχνουμε στο πλαίσιο του ETS μέχρι το 2030 ε, ε, είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα βοηθήσει στην καινοτομία ακόμη και αν ληφθούν τα μέτρα. Ε, ακόμη και αν δεν μας νοιάζει η εφαρμογή των παρεσίων θα δούμε κατακαιρματισμό ουσιαστικά της εφαρμογής από, κράτος μέλος, από το ένα στο άλλο και ήθελα να δούμε τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό Όσον αφορά τώρα τη μακροπρόθεσμη ατζέντα για το 2050, επίση σημαντική, στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να δώσουν ε, μακροπρόθεσμου ε, οδικού χάρτε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό που είναι όλο και πιο σημαντικό είναι αυτοί οι οδικοί χάρτε να βασιστούν ε, στον προπολογισμό άνθρακα. Η εμπίστηση αναφέρεται σε συγκεκριμένο προπολογισμό άνθρακα που θα είναι διαθέσιμος. Η Κομισιόν στη δική της ανάλυση τώρα θα δώσει πληροφορίες προς τα κράτη-μέλη ποιος θα είναι ο προπολογισμό άνθρακα εντός του οποίου θα πρέπει να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτή θα είναι μια σημαντική συζήτηση μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ελπίζω οι Κομισιόν να δώσουν πληροφορίες τέτοιες για αυτόν τον προπολογισμό άνθρακα, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τα κράτη-μέλη τα μακροχρόνια σχέδιά τους. Ήθελα να πείτε την άποψή σα. Τέλο για την αεροπλοεία. Μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχει καταλήξει η Κομισιόν σε αυτή την ε, ε, ασαφή πρόταση της, ε, του παγώματος των δραστηριοτήτων του Stop the Clock. Δεν φαίνεται να έχει κάποια συγκεκριμένη καταλήξη και δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν το έκανε. Και μετά γιατί προτείνει η Κομισιόν από το 2021 δεδομένου ότι θα εφαρμοστεί η Κορσία. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει αλλά θα εφαρμοστεί η Κορσία. Γιατί δεν προτείνουμε κάτι για να είμαστε βέβαιοι ότι η Κορσία θα συμπεριληφθεί στο ETS ώστε η ευρωπαϊκή προσέγγιση του ETS να είναι η μετάφραση του Κορσία στην ευρωπαϊκή αεροπλοεία ώστε να έχει νόημα. Αυτό ήθελα να ακούσω ως άποψη από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του EFDD, κυρία Εύη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ. Και εμεί το κίνημα των πέντε αστέρων, ναι, ήμασταν ιδιαίτερα επικριτικοί για το ETS. από το σκεπτικό που άκουσα να διατυπώνεται. Χαίρομαι που ακούω και διάφορες φωνές ε, επικριτικές ε, σε σχέση με αυτό το εργαλείο, το οποίο πράγματι δεν φέρνει αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία, οι μόνες δράσεις που πραγματικά μείωσαν τις εκπομπές πέραν των ε, μειώσεων λόγω του κλεισίματος διαφορών βιομηχανιών και, ε, και λόγω της μείωσης της παραγωγής αφορούν αποκλειστικά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τα μέτρα ανάπτυξης ε, και διάδοσης των ενωσιμών πηγών ενέργειας δεν οφείλονται στην οδηγία ETS. Ε ε, τίποτα δεν φαίνεται να οφείλεται στο ETS. Ε Ωστόσο, στο κείμενο που συμφωνήθηκε στο Κοινοβούλιο, εκφράζεται μια ανησυχία, υπενθυμίζω, όσον αφορά το γεγονό ότι οι πολιτικές κλίματος και ενέργειας επηρεάζουν την αγορά του διοξιδίου του άνθρακα. Εξακολουθούμε δηλαδή να μιλάμε για αγορά διοξιδίου του άνθρακα. Εξακολουθούμε να θέλουμε να την προστατέψουμε. Συνεχίζουμε προφανώς να θέλουμε να θυσιάσουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο βωμό της κερδοσκοπίας Και αυτό ε, το διαπιστώνουμε εκ των πραγμάτων ε, λόγω της, ε, βλέποντας τις ανυπαρκείς φιλοδοξίες του χειμερινού πακέτου για την ενέργεια. Δεν θεωρείτε κύριε Επιτρόπε ότι έχει έρθει η ώρα να αντιστρέψουμε την τάση και τις προτεραιότητες να κάνουμε πιο φιλόδοξους τους σημερινούς μετριοπαθείς στόχους για ε, την εξοικονόμηση ενέργεια και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αντί, κύριε Κανιέτα, να διατηρούμε ένα μοντέλο που, όπω γνωρίζουμε από την εμπειρία μα ε, στην πραγματικότητα και με τα στοιχεία στα χέρια μα, ότι δεν έχει λειτουργήσει. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε πορεία. Δεν φοβάστε ότι θα είναι αργά όταν θα αντιληφθούμε ότι χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Ε, Θα είναι πολύ αργά όταν χάσουμε την ευκαιρία. Κύριε Ντοχνάνο, <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η πρώτη μου ερώτηση αφορά το σεβασμό των στόχων μείωσης ε, των αριών του θερμοκηπίου. Με την έγκριση της συμφωνίας ΣΕΤΑ με τον Καναδά, η απελευθέρωση του εμπορίου Ευρώπης-Αμερικής μηχανικά θα οδηγήσει στην αύξηση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Χειρότερα ακόμα, οι δικοί μας αγρότες θα έρθουν αντιμέτωποι με ε, αγρότες του Καναδά που έχουν 35% χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Και επίσης οι τόποι παραγωγής έχουν την τάση να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τους τόπους κατανάλωσης των τροφίμων. Οπότε έχουμε μεγάλη ε, αύξηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ερώτηση λοιπόν για να σεβαστείτε τους πάρα πολύ ε, φιλόδοξους στόχους σας. Μείωση πάνω από 40% για το 2030 των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 90. Σε ποιον τομέα της οικοδομίας μας θα ζητήσετε να γίνουν ε, μεγαλύτερες προσπάθειες για να αντισταθμιστεί η επίπτωση της συμφωνίας ΣΕΤ. Δεύτερη ερώτηση, διαχείριση των δασών και εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιλίου 2016 ασχολούνται με την καταμέτρηση των εκπομπών από ε, το ξύλο που χρησιμοποιείται ε, ως καυσόξυλο. Αλλά δεν είναι αυτός ε, ο βασικός λόγος, η βασική πηγή εκπομπών. Έχουμε πρώτα τις μεταφορές, μετά τη βιομηχανία, μετά το μαζούτ και μετά το αέριο. Και στη συνέχεια τα καυσόξυλα. Ε, επίσης ε, τα δάση δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα και ανανεώνουν τα δέντρα. Και πολλά δέντρα επίσης ε, δεσμεύουν τα αιωρούμενα σωματίδια που προκύπτουν από την αποτέφρωση ή από την κάψη των ξύλων. Άρα εσείς αναγνωρίζετε ότι το ξύλο είναι σχετικά η φόρος πηγή ε, ε, ενέργειας ή μήπως θέλετε ε, κάποια στιγμή να απαγορευτεί αυτή η πηγή ενέργειας για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπο για τις απαντήσεις Ευχαριστώ πολύ Επίτροπος για να απαντήσει. Παρακαλώ. Με χαρά θα σας ακούσουμε. Βεβαίω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτάς οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών ή και τόσο όσα στο Συμβούλιο και εκεί αλλά και εδώ ήταν τα πράγματα δύσκολα και περίπλοκα. όπως και το θέμα είναι περιπεπλεγμένο. Και εσείς έχετε επικρίνει το σύστημα ότι δεν έχει καλές επιδόσεις κλπ. Αλλά για πρώτη φορά συνειδητοποίησα τις προάλλες κατά τη συζήτηση ότι έχει και κάποιες φιλοδοξίες σχετικά το Συμβούλιο. Τα είχαμε συζητήσει εκεί, όπου και εκεί είχαμε τις διαρροές. Άρα έπρεπε να υπάρξει προσοχή, αξιόλογη συζήτηση και υπάρχει τώρα το πλαίσιο για συμφωνία. Τώρα πόσο καλές επιδόσεις θα έχει μετά το σύστημα και εσείς επικρίνετε επομένω, ε, είναι και θέμα εθνικών μέτρων. Σύστημα που να έχει σχέση με τις αγορές, με τιμολογική πολιτική, φορολογική πολιτική, μα δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αγορά. Την αγορά του άνθρακα και οπότε τώρα υπάρχει κάποια δυνατότητα. Γιατί για πρώτη φορά οι θέσει ειδικέ σα και το Συμβούλιο δεν αφήστανται τόσο πολύ, οπότε μπορούμε τώρα κάτι να κάνουμε. Όλοι είναι απεσιόδοξοι. Από το 1,74 πάμε στο 2,2 ακόμα το 2,4 ως οροφή. Και αυτό δεν είναι δεκάρες. είναι πολύ σημαντικό. Οπότε βελτιώνουμε σιγά σιγά το σύστημα στη λειτουργία του. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο. Η προϊστορία δεν είναι τόσο ρόδινη. Γι' αυτό και έχουμε κάνει διαδοχικές βελτιώσεις. Όμως ήρθε η ώρα να επιφέρουμε περισσότερες μεταβολέ. και να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε Κύριε Λίζε, είπατε για την κατανομή τη ευθύνη των προσπαθειών και τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Καλά, αυτό ισχύει για όλα τα θέματα. Έχουν προστεί επικρίσει και εγώ πολλού έξι μόνο ότι δεν κάνω όσα μπορώ. Όχι. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει και κάνω ό,τι μπορώ. Όσο πιο φιλόδοξο μπορώ να είμαι. Και για τη διαδικασία των συμβασμών και για τον τριμερή διάλογο. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν συμφωνούσαν με την γενικότερη προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να ένα συμβιβασμό και να συσπηρώσει όσο γίνεται περισσότερους. Άρα ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πολλά και σημαντικά είπατε. Είπατε για τις μεταφορές και για τα λόμπια. Σίγουρα για τα οχήματα, το να καθορίσουμε του στόχου δεν είναι κάτι το εύκολο. Σαν αφορά εκπομπέ, εδώ και μισή χρόνια καταβάλουμε προσπάθειε, έχουμε ένα σωρό μελέτε κλπ. Προσπαθούμε με μελέτε επιπτώσεων. Αλλά έχει καταστεί σαφέ ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα είναι διαφορετική από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Γιατί ακριβώ τώρα θα κάνουμε αυτή την στροφή από το NDC στο WLTP και με τις νέες προτάσεις πρέπει να δούμε εντατικά και επιγόντως τι θα κάνουμε με την ηλεκτρική κινητικότητα. Μας είπατε και για τα λόμπι, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι κατάλαβα, στα πλαίσια της αυτοκινητοβιομηχανίας η εξέλιξη τέτοιων ε, οχημάτων προχωράει. Βέβαια, τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτε. Να δούμε τι τεχνικέ εξελίξει θα έχουμε. Όμω θα πρέπει να στηρίξουμε αυτέ τι προσπάθειε και στο μέλλον. Θα πρέπει να ενεργήσουμε και νομοθετικά. Και όσον αφορά τη φόρτιση. Αν δεν υπάρχει υποδομή για φόρτιση, τι κινητικότητα να έχουμε. Γι' αυτό είδατε ότι έχουμε τη σχετική οδηγία, τη σχετική δέσμη για το clean energy, για τους Ευρωπαίους λοιπά Και για τις μπαταρίες είπαμε, γιατί για να είναι η κινητικότητα αυτή ε, ε, ελκυστική είναι και θέμα τιμής. Είναι και θέμα βεληνικούς των μπαταριών. Άρα, θα προτείνουμε στόχους, αλλά θα παίζει σημαντικό ρόλο στη δέσμη μέτρων η κινητικότητα. Και θέλουμε να πετύχει δέσμη μέτρων. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς παράγεται η σχετική ενέργεια για την ηλεκτρική κινητικότητα. Άλλος ρώτησε για τα ανανεώσιμα και ότι δεν είμαστε φιλόδοξοι στις προτάσεις μας και ότι χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι. Ε, βέβαια, αν έχετε δεσμευτικούς στόχους, ε, αν κάποια κυβέρνηση δεν πετύχει τους στόχους, τον, το προσάγουμε στο δικαστήριο. Τώρα όμως, είναι διαφορετικό το σύστημα. Για πρώτη φορά έχουμε αυτά τα ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα. Περιλαμβάνει και το κλίμα και τα συζητήσαμε μια που οι πρακτικέ συνθήκε στα κράτη-μέλη είναι στο καθένα διαφορετικά. Εσεί μα μιλήσατε για την Ιρλανδία, μα είναι σαφέ ότι οι προποθέσει για τα ανανεώσιμα δεν είναι ίδιε από χώρα σε χώρα. Άρα θα πρέπει να γίνει κουβέντα για την ευελιξία. Και σε αυτή έχουμε και κάποιε κυβερνήσει με τις οποίες ελπίζουμε ότι τελικά θα τα βρούμε. Θα γεφυρωθεί διαφορές και βέβαια αν δεν τα βρούμε θα μπορεί το Κοινοβουλίο να τροποποιήσει τον κανονισμό. Οπότε θέλουμε δεσμευτικούς στόχους που να είναι επιτρέψιμοι. Αλλιώς χωρίς ισχυρή διακυβέρνηση δεν γίνεται. Γι' αυτό έχουμε και αφετηρία τους παλαιότερους κανόνες για την διακυβέρνηση. Και έτσι προχωρήσαμε στην καθαρή για τους Ευρωπαίους σε όλο αυτό το πακέτο. Και ελπίζω το Κοινοβούλιο πρόκειται να βελτιώσει τις προτάσεις μας. Μας πέτυχε για τα νησιά. Να έχουμε και μια σχετική πρωτοβουλία. Θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα συζητήσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία. Τώρα το επεξεργαζόμαστε για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων, την διασυνδεσιμότητα και έτσι να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε αυτό το μέτωπο. Όμως υπάρχει πρόβλημα στα νησιά. Έχει ο κόσμος εκεί πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσουμε για το πώς θα αναπτύξουν ενεργειακή ένωση. Θα με δώσει προτεραιότητα στο κεφάλι αυτό στο παρελθόν και στο μέλλον. Στη συνέχεια. Σε σχέση με αυτά που ρώτησε Κύριε Κέρλινγκ, για τα βιοκαύσιμα. Τα προηγμένα. Έχουμε ελάχιστα ποσοστά και κάνουμε και άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μειώνουμε ε, το βάρος των ε, βιοκαυσίμων που παράγονται από φυτά που μπορούν να παράγουν και τρόφιμα. Βεβαίως αυτό είναι μια νομοθεσία που θα χρειαστεί χρόνια, δεν είναι του παρόντο, αλλά γίνεται προσπάθεια αυτό το καιρό στα βιοκαύσιμα. Υπάρχουν πολλές καινοτομίε και εμείς θα το υποστηρίξουμε με το Horizon 2020 ε, και άλλα ερευνητικά προγράμματα. Βεβαίως, ε, οι ορισμοί στις προτάσεις μας μπορεί να είναι πολύ ασαφείς ή πιο συγκεκριμένοι, θα το δει αυτό το κοινοβούλιο, θα το επεξεργαστεί. Αλλά προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει στην πρότασή της. Αναφερθήκατε στη διαφάνεια στον ΑΙΚΑΟ. Μα τα συζητούμε αυτά τα θέματα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε ε, ε, ενεχόμενο μέρος της Συμφωνία των Παρισίων, της Κλιματικής ε, Συμφωνία ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματευόμαστε με διαφάνεια, ενημερώνουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Διότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να συμφωνήσουμε στον ΑΕΚΑΟ κανόνες για τεχνικά στοιχεία για το νέο σύστημα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ακαιρεότητα του συστήματος. Όλοι οι κανόνες για την παρακολούθηση, την αναφορά, τις επαληθεύσεις κτλ. Ε, όλα αυτά ε, να καταμετρώνται και να υπάρχει μια ε, λογιστική ας πούμε, καταγραφή των εκπομπών με τρόπο διαφανή και υπόλογο και αξιόπιστο και για τα βιοκαύσιμα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ποιες είναι οι μονάδες εκπομπών που είναι επιλέξιμες για τη συμμόρφωση. Γιατί υπάρχει ένα στοιχείο προσθετικότητας και υπάρχουν προβλήματα με τα διεθνή ε, ανταλλάγματα, εξισορρόπηση, υπάρχουν ε, διεθνείς ε, υποχρεώσεις από τη Συμφωνία των Παρισιών για να μην υπάρχουν διπλές αξιώσεις και διπλές αποζημιώσεις. Και η Κόρσια είναι ένα σύστημα ε, πραγματικά ε, που πρέπει να δοκιμαστεί στην πράξη. κατά όλα αυτά που ζητάτε για τη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία. Αυτά θα τα δούμε στην Επιτροπή Μεταφορών για να είναι το Κοινοβούλιο ενήμερο για τις αλλαγές ή τη συντημορία των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να έρθουν στο Κοινοβούλιο και να συζητηθούν. Ο κύριος Γκερμπράντι ε, έκανε μια από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις και περίπλοκες. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Ε, έχουμε μια συμφωνία διαπραγματευτή. Αρχίσαμε ε, όλα τα νομοθετικά αυτά βήματα να κάνουμε με την εργαλειοθήκη, τι είναι νομοθεσία, την συμφωνία, αλλά τα ξέρει αυτά η κοινή γνώμη. στις δημοσκοπήσεις ε, λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι η κλιματική πολιτική είναι σημαντική για εκείνους. Αλλά ξέρουν τι χρειάζεται να γίνει για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Θα είναι αυτό ένα θέμα που θα κυριαρχήσει στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ. Τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και είναι ένας από τους τομείς πολιτικής που μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα αν θέλουμε μια πιο φιλόδοξη Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λανσάρει τέτοιε συζητήσει στα κράτη-μέλη και με ζητήματα για το κλίμα. δείτε τη Λευκή Βίβλο, η κλιματική πολιτική είναι μία από τις δράσεις, όπου λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει κτλ. Ορισμένοι λέγουν ότι έχουμε λες, μικρή πρόοδο, αλλά θα πρέπει να το μάθει και ο κόσμος. Θυμάστε τις περασμένες ευρωεκλογέ. Ποιο θέμα κυριάρχησε κάποια στοιχεία του eco design, οικολογικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή ποιο θα είναι ο σχεδιασμό οικολογικό των διαφόρων συσκευών τη τοστιέρα, τη φρυγανιέρα κτλ. Αυτό μα μάρανε. Και πριν το 2020 ε, θα πρέπει να βάζουμε τους νέους στόχους και το 2020 23 να έχουμε πιο φιλόδοξες προτάσεις. Τώρα έχουμε και τη μόδα τον όρο το Spitzenkandidat που είναι επικεφαλή του ψηφοδελτίου και σπρώχνονται διάφοροι να τεθούν επικεφαλή. Και για ρωτήστε του τι θα κάνουν για το κλίμα. Φέτος θα έχουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση, αλλά στι ευρωεκλογέ θα είναι ακόμα πιο σημαντική βασικά τα προγράμματα και οι υποψήφοι. Ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο ή ποια θα είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιε πολιτικέ θέλει να επικεντρωθεί. Αυτό είναι η σημαντικότερη πρόκληση. Και από εκεί και πέρα θα ξαναπούμε. Ε, συμφωνώ πολύ κύριε Γκερμπράντη, Γιατί ο κόσμο δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Πηγαίνω σε διάφορα κράτη-μέλη και η συζήτηση γίνεται αμυγό εθνική. Όπω είπε η κυρία Τόρε Μαρτίνεθ. Αυτά τα θέματα είναι εθνική πολιτική, δεν είναι η παγκόσμια πρόκληση και πώς θα αντιμετωπίσουμε με φιλοδοξία τα προβλήματα και ποια θα είναι η δράση μας. Και είναι μια καλή ευκαιρία αυτή κύριε Κεμπράντη τώρα με τα εθνικά ολοκληρωμένα προγράμματα, ε, τα ενεργειακά και τα κλιματικά των κρατών μελών, τα επιχειρησιακά σχέδια, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν για μια δεκαετία ένα πρόγραμμα χωρίς να ανοίξει μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για την κλιματική υπόθεση και χωρίς να συζητήσει με τους ενδιαφερομένους και τους ενεχομένους. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει όταν δρομολογηθεί αυτή η συζήτηση. Το 2018 θα κάνουμε προτάσεις και το 2019 και έχουμε και στρατηγική για χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν τα προγράμματά τους για μια δεκαετία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα πρέπει να το συζητήσουμε στις 27 πλέον και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η σωστή κατάλληλη συγκυρία, γιατί χρειάζεσαι υποστήριξη από τους πολίτες για να εφαρμόσεις κάποιες πολιτικές. Άρα η συζήτηση αυτή θα ανοίξει το 2018 και θα κλείσει στις ευρωεκλογές και όλα τα μανιφέστα των κομμάτων. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω κι εγώ Γιατί ε, ξέρω ότι πολλές πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο ε, το έχουν αυτό το θέμα προτεραιότητα. Και θα υπάρξουν και πολιτικά κόμματα που θα το αναδείξουν. Και θα γίνει και συζήτηση στο debate μεταξύ των υποψηφίων. Εκεί να δείτε ενδιαφέρον που θα έχει συζήτηση αυτή. Συναρπαστική θα είναι. Mm. Για το θέμα με τις ΗΠΑ που ρωτήσατε, είναι πρόωρο ακόμα. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τι στάση θα κρατήσουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ε, όσον αφορά την αναγνώριση των ανθρωπογενών ε, παραγόντων που οδηγούν στο ε, κλιματική αλλαγή ο σχετικός υπεύθυνο τη ΕΙΠΑ θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο έχω μειώσει τον προπολογισμό 20-30% αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη για το προς τα που θα κινηθούν ένα πράγμα είναι σαφές. Η δέσμευση του Πρόεδρου Ομπάμα δεν θα υπάρξει. Ούτε η δέσμευση του κυρίου Κέρι. Δεν έχουν ε, ορίσει ειδικό απεσταλμένο για το κλίμα. Που θα είναι ομολογός μου, ε, για να το πω έτσι. Συζητώ με το State Department, με το Λευκό Οίκο. Αλλά οι ομάδες αυτές δεν έχουν ακόμα συσταθεί. Και οι προηγούμενες ε, ομάδες ε, έχουν εξαφανιστεί. Ε, απομακρύνθηκαν. Οπότε μας είναι άγνωστο το μέλλον. Θα πρέπει να κάνουμε επαφές μόλις διοριστούν τα σχετικά πρόσωπα και ξέρουμε ότι ο ρόλος του Λευκού Οίκου και του State Department θα είναι σημαντικός. Ε, θα δούμε πρώτα απ' όλα αφού ε, ε, διοριστούν όλοι οι αρμόδιοι. Θα δοκιμάσουμε όμως τα πράγματα στη Βόνη όπου σύντομα θα συζητήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η στάση τους. Και έχουμε και την ΚΟΠ, την ΚΟΠ23 στη Βόνη. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Να θυμάστε ότι οι ΙΠΑ αποχώρησαν από το πρωτόκολλο του και ότο μια φορά και χρειάστηκε πολύ καιρό μέχρι να ξανέρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Τώρα θα αναλύσουν τι έχει συμβεί σίγουρα και θα δράσουν ανάλογα. Τώρα με ρωτήσετε για την Κίνα, ναι είναι βέβαιο. Σε μια-δυο εβδομάδε θα μεταβώ στην Κίνα, εγώ, για να συζητήσουμε τις αγορές άνθρακα και την κλιματική πολιτική και είμαι βέβαιος ότι στη διασκέψη κορυφής θα συζητήσουμε πρωτίστως τη δράση της Κίνας για το κλίμα. Είναι σαφές ότι οι διεθνείς συνομιλίες ε, για το κλίμα είναι διαφοροποιημένες, ε, είναι ποικιλόμορφες, ε, δεν είναι υποχρεωτικά να συμμετέχει. Οπότε αν οι δεν θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ηγηθεί κάποιο άλλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ε, πολλά πράγματα ήδη. Έχει ήδη κλιματική διπλωματία, έχει όλες τις επαφές που χρειάζεται για την υπεράσπιση και την εφαρμογή των Σύμφωνων των Παρισίων. Και αυτό πιστεύω αποτελεί τεράστια ευκαιρία για μας. Η κυρία Τόρες Μαρτίνες που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή μαζί μου, θα ήθελα να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, για τις διασυνδέσεις. Αν δείτε τι υποδομές έχουμε χρηματοδοτήσει. Τι έχει υποστηρίξει η Κομισιόν. Έχουμε καταπολεμήσει την απομόνωση της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης μέσω συστηματών διασύνδεσης ώστε οι χώρες αυτές να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες ροές παροχής φυσικού αερίου. Δεν μιλάμε για τεράστια έργα διασύνδεσης, μιλάμε για υποστήριξη μικρών έργων στη Βουλγαρία, στη Σερβία, Βουλγαρία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία έχουν διασυνδεθεί και εμείς το έχουμε υποστηρίξει. Δεν κάνουμε μεγάλες, ε, ε, μεγάλους αγωγούς. Μόνο αυτό του νότιου διαδρόμου ε, από το Ιζερμπετζάν μέχρι την Ιταλία έχει υποστηριχθεί που αποτελεί κυρίως ιδιωτική επένδυση αλλά και υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θεμελιώδη σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ε, λέγατε τι γίνεται με το φυσικό αέριο και ποιο πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αν δείτε τις εκτιμήσεις μας όσον αφορά την κατανάλωση ε, του φυσικού αερίου μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί ε, και τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά ποια είναι πιο καθαρή το φυσικό αέριο. Οπότε θα χρειαστεί μέχρι το 2030 από 380 έως 450 BCF ε, ε, φυσικό αέριο. Είναι κάτι που δεν θα εξαφανιστεί, θα, είναι μια ανάγκη υπαρκτή. Εμείς χρηματοδοτούμε υποδομές για να μην μένουν ακίνητα, για να μένουν αχρηστές, αναλύουμε κατά πόσο θα ε, χρησιμεύουν. Τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Συνδέουμε χώρες της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης μεταξύ τους και με τα μεγάλα δίκτυα φυσικού αερίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ευφυής πολιτική για την ασφαλή του εφοδιασμού και για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Με κατηγορείτε... Θα πέρασω στα ισπανικά, συγγνώμη. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Συνεργικής Πολιτικής ενσωματώθηκε σε κάποιο νομοθέτημα το δικαίωμα των καταναλωτών να παράγουν οι ίδιοι την ενεργειά τους και να την πολλούν, να την αποθηκεύουν και το κόστος να μην είναι υπέροχο. Το πρότεινα εγώ, ταπεινά. Κοινοτική νομοθεσία η οποία πρέπει να τηρείται και αν κάποια κυβέρνηση τη Α τη Β χώρα, όταν ισχύσει αυτή η νομοθεσία δεν την τηρήσει ε, τότε θα ε, το στέλνουμε στο δικαστήριο για διαδικασία παραβάση. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό το δίκαιο. Και δεν λέω μόνο για τις μικρές, θα ξεκινήσουμε από τους μεγάλους, τις μεγάλες χώρες. Συνέχεια, κάθε μήνα θα το κάνουμε αυτό. Εμείς, οι επίτροποι, δεν θεωρούμε ότι ανήκουμε σε κάποιο κόμμα ή ότι εφαρμόζουμε εθνική πολιτική. Ο κύριος Έκχαρτ έβαλε μια σειρά ερωτήσεων σε σχέση με την κοινή αγορά. θα προσπαθούσαν να έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά που να αποδίδει και να μπορεί να συνδέεται και με τις υπόλοιπε αγορές σε όλο τον κόσμο. Ε, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις χώρες να αναπτύξουν αγορές άνθρακα, διεθνείς πρωτοβουλίες, διμερείς όπως με την Κίνα και έχουμε και αυτή την πολύ μεγάλη διάσκεψη σχετικά για να αναπτυχθεί ένα σύστημα Σίγουρα μπορούμε να έχουμε επιπλέον προσπάθειες των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία εδώ αλλά και στο Συμβούλιο να κλειστεί η συμφωνία που θα φέρει ουσιαστική βελτίωση από όσα προτείνουμε τον Οκτώβριο του 2014 αυτές τις ε, λειτουργικές ρυθμίσεις για το σύστημα εκπομπών. Είμαι βέβαιος, έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, ο Σεκάτ μας είπε και για τον προπολογισμό σχετικό με τον άνθρακα, ξέρετε, σε σχέση με το κλίμα και τα σχέδια κειμένου προτάσεις που υπάρχουν από τις κυβερνήσεις, υπάρχει προβληματική για τη διακυβέρνηση, να δούμε πώς θα ε, τι, τη μορφή θέλουν αυτά τα εθνικά προγράμματα, αλλά εμείς εμένουμε σε αρχή μας πρόταση. Και αυτό το οποίο θα πάμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει η ρύθμιση, η ρύθμιση του 18 στα πλαίσια της στρατηγικής ε, μείωσης του άνθρακα, περικοπής του άνθρακα. Και αν γίνει σχετική ανάλυση και από κοινωνικής πλευρά, όλα όλα θα τα λάβουμε υπόψη να δούμε πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική, η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από ορόσημα, από στόχους, από ποσοστά, από εκατομμύρια τόνους. Στρατηγική πάει να πει ανάλυση των επιπτώσεων οικονομικών, κοινωνικών, για κάθε κλάδο της οικονομίας. Χρειάζονται βιομηχανικές μεταρρυθμίσεις, μετασχηματισμοί και η γνώμη μου θα είναι ό,τι πιο δύσκολο έχει να κάνει αυτή τη θητεία η Κομισιόν. Αυτή η στρατηγία για τον άνθρωπο Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Εύκολο είναι να βάζει κανεί στόχου και χρονοδιαγράμματα και αυτά. Όμω θα πρέπει κανεί να κλείσει εγκαταστάσει. Θα πρέπει να, ρυθμίζει, να αλλάζει. τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Όμω με ένα θετικό τόνο κλείνουμε ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να επιδείξουμε δηλαδή την πολιτική βούληση να τα βρούμε. Οπότε γι' αυτό και την επόμενη διετία με αυτό θα ασχοληθώ, με αυτή τη στρατηγική. Χέρι-χέρι με εσά. Τέτοια προσέγγιση θέλω. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ποιος το είπε, η κυρία Α, τώρα Μαρτίνας, είπε είπαμε για 80-90% έχουμε τους στόχους για τον άνθρακα τους έχουμε τάξει και πριν τη διάσκεψη των Παρισίων ε, τώρα θα πρέπει να έχουμε δύο των άνθρακα υπόψη στο Παρίσι να δούμε τι θα πετύχουμε πότε τα πράγματα είναι διαφορετικά να άλλη στατική τώρα διαφορετική δεν πάμε για 80-90 ή πάμε για παραπάνω και αυτά θα είναι εκπεφρασμένα όχι μόνο με στόχους αλλά με επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές. Δύσκολο. Τι άλλο έχουμε εδώ. Α, για, να σταματήσουμε το ρολόι για την αεροπλοεία και το κόρσια. Αυτό ακόμα εκρεμεί αλλά εξαρτάται ε, από το πώς θα δουλέψει το σύστημα κόρση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να έχουμε φιλόδοξους στόχους έρευνας στον Ναϊκά, με ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες μας. Αλλά Φέραμε την πρόταση αυτή στο Κοινοβούλιο, μπορεί το Κοινοβούλιο να την τροποποιήσει κατά το δοκούν και από εκεί και πέρα. Το μόνο που ζητούμε είναι ταχύ αντίδραση του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να ε, προλάβουμε ε, τις προθεσμίες στον ΑΕΚΑΟ. Το θέμα το γνωρίζουμε όλοι. Ξέρουμε όλες τις επιπτώσεις, όλες τις αποχρώσεις στην αεροπλοεία. Ε, ελπίζω να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα με μια λογική ταχύτητα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρω ότι θέλετε όλοι να κάνετε ερωτήσεις προς τον Επιτροπό. Έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε μία ερώτηση. ώστε να προλάβει και ο Επιτροπός να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της ε, Επιτροπής, τον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ. Γνωρίζω τους χρονικούς περιορισμούς που έχουμε. Μια απλή ερώτηση λοιπόν στον Επίτροπο για τον επιμερισμό προσπαθειών. Ξέρετε, Επίτροπε, στην πρόταση της Κομισιόν τα αρχικά στοιχεία για κάθε χώρα είναι τα τελικά στοιχεία της προηγούμενης περίοδου. Οπότε οι χώρες που έκαναν προσπάθειες, τις μεγαλύτερες προσπάθειες και που δεσμεύτηκαν για την επίτευξη στόχων πιο φιλόδοξων από τους target, τελικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην επόμενη περίοδο. Διότι κατέβαλαν τις προσπάθειες και περισσότερες αρχικά Πώς θα διορθώσει η Κομισιόν ε, αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζει η πρόταση και που θέτει σε δύσκολη θέση κάποιες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Όταν η αυτόνομη παραγωγή ενέργειας ε, όλο ένα ε, αυξάνεται και υπάρχουν όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα προβλήματα διαχείρισης των δικτύων είναι όλο περίπλοκα δεν είναι λοιπόν ε, αρνητικό το να, ε, να επηρεάζουμε με αυτόν τον τρόπο την εκμετάλλευση, τα δίκτυα εκμετάλλευσης ενέργειας. Έχω μία ερώτηση. Είμαστε εδώ πόση ώρα, μία ώρα και 15 λεπτά. Πέντε ερωτήσεις έχουμε ακούσει και πέντε απαντήσεις. Τώρα θα επικρίνω εν μέρη τον ε, Επίτροπο, ο δίνει ε, μεγάλες απαντήσεις. Είμαστε όλοι πολιτικοί εδώ, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Μιλάτε όσο μπορείτε περισσότερο και σα κάνουν λιγότερε ερωτήσει. Αυτό δεν είναι πολύ δημοκρατικό. Αλλά η βασική μου κριτική είναι, κυρία Πρόεδρε, υποτίθεται ότι προεδρεύετε την Επίτροπη. Δεν την ε, προεδρεύετε, απλά κάθεστε και δεν προεδρεύετε. Πρέπει να ελέγξετε τα πράγματα. Εδώ είναι η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να τον ελέγξετε. Τον έχετε καλέσει εδώ και πρέπει να τον ελέγχετε. Και αυτός ε, έχει ε, καταλάβει όλη τη συνεδρίαση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είτε θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθείτε ως πρόεδρος ή να σταματήσετε να προεδρεύετε. Δεν έχει νόημα να κάνω ερώτηση. Είναι χάσιμο χρόνο γιατί μέχρι να ρωτήσουν όλοι τις ερωτήσεις τους ε, θα πάει 8.30, δεν θα έχουμε μεταφραστές, οπότε... Είναι απαράδεκτο. Εγώ θα αναχωρήσω και παρακαλώ βελτιώστε τις ικανότητες σας, Πρόεδρε, στις συνεδρίες σας. Κύριε Μπέρνου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυσνιεύσκα. Συγγνώμη, έχω μία λίστα ομιλητών που μου δόθηκε από τη γραμματεία. Που δόθηκε στη γραμματεία από τους συντονιστές, εκτός μικροφώνου, κύριε Πρόεδρος. Ο πρώτο ήταν ο κ. Μπράνεν και τώρα πάω στο ΕΣΥΑΡ. η κυρία Βυσνιεύσκα. Τι να πω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, στην τελευταία συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος το Συμβούλιο θέτησε μια θέση για τη μεταρρύθμιση του ΙΤΕΣ. Εννέα χώρε,. Ε, προτάθηκαν και ήθελα να μάθω αν ε, ο ε, συμβασμός Διανίνα ε, ισχύει ακόμα και αν η Επιτροπή ελέγχει ακόμα αυτή την πολιτική και είναι σε θέση να αξιολογήσει τις συνεπίες της. Η επιβολή πολιτικών θεωρείται είναι καλή λύση. Ευχαριστούμε. Ε, το κόμμα σας, ε, το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία, και ήσασταν, έχετε διατελέσει υπουργό και γεωργίας και υπουργό περιβάλλοντος. Έχει στηρίξει κάτι που κατά την άποψή μας είναι αμφισβητήσιμο. Η παράταση της χρήσιμης ζωής σε 60 χρόνια ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων, πυρηνικών εργοστασίων που είναι ένα, ε, ε, συγκεκριμένο ένα από τα δέκα αρχαιότερα παγκοσμίω. Και αυτό γίνεται και άσκοπα και αυτό είναι το χειρότερο. Στην Καρόνια, στην Ισπανία, ε, αυτός ο σταθμός παράγει μόλις το 1% ε, της ηλεκτρικής ενέργειας που εμείς καταναλώνουμε. Και ρωτώ κύριε Κανιέτη σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Ευρώπη και η Ισπανία έχουν υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ε, οπότε η πυρηνική ενέργεια δεν θεωρείται υποστηρικτική προς τις ανανεώσιμε γιατί δεν είναι ευέλικτη. Επιμένετε εσείς να διατηρηθεί η πυρηνική ενέργεια όπως κάνει το κόμμα Και επόμενη ερώτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις ε, πυρηνικούς αντιδραστήρες στον κόσμο θα είναι σε λειτουργία πάνω από 40 χρόνια το 2020. Μήπως θα θεωρηθεί προηγούμενο να ανοίξει ένας τέτοιος πυρηνικός σταθμός στην Ισπανία για να παρατηθεί η διάρκεια ζωής αυτών των πυρηνικών ε, καταστάσεων που είναι και επικίνδυνες εκτός του ότι είναι ε, υπέργυρες. Κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σύμφωνα με την αξιολόγησή μα, ε, υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα τόσο για το 2025 όσο και το 2050. Και αυτό είναι ο καλύτερο καλύτερος τρόπο είναι το να υιοθετήσουμε τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σα εκτίμηση. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε ε, πληροφορίες, οπότε σας ξαναρωτώ ρητά. Η Κομισιόν και εσείς θα κάνετε κάποια πρόταση για το 2025 και το 2030 με σχετικούς στόχους για τα δύο αυτά έτη επίπεδου τέτοιου που να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσει της Συμφωνίας των Πορυσίων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για τους καταναλωτές ε, όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των οχημάτων. Επιπλέον θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε σήμερα να το υποσχεθείτε, μιλήσατε για κύκλους δοκιμών ότι η πρότασή σας θα θέσει νέα όρια διευθυντήτου του ανθράκα βάσει πραγματικών ε, τεστ ε, οδήγησης. Η Κομισιόν ε, τι θα κάνει με τα πρότυπα των βαρέων οχημάτων. Θα βάλει ε, θα δημιουργήσει και εκεί νέα στάνταρ. Ευχαριστώ κυρία Καμπεζόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ε, να εκφράσω τη δυσφορία μου στην αρχή για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται εδώ η συζήτηση. Δεν μπόρεσαν οι βουλευτές να ρωτήσουν, να μιλήσουν καθόλου. Εν πάση περίπτωση, παρόλα αυτά θα κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορα τις ερωτήσεις μου για να μιλήσει και άλλος συνάδελφος. Διατηρώ αμφιβολίες, πρέπει να σας πω, για την τήρηση των στόχων του συμφωνίας του ε, Παρισιού 27% ανανεώσιμες το πέμπτο ε, πακέτο κάτω από 30% που το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει, 6,8% για τις μεταφορές ανανεώσιμες, ουσιαστικά στο 6% είμαστε ήδη. Άρα ποιος είναι ο στόχος που θα δώσει κίνητρα να ανταποκριθούμε. Που μας τα προτείνεται και μας τα παρουσιάζεται ως τα βασικότερα μέτρα που ενδιαφέρεται και ο κλάδος. 30% ενεργειακή απόδοση και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, είναι επαρκέ γιατί βάζει και ένα μέτρο ευελιξίας. Ε, Όπω ρώτησε και η κυρία Μίρια Μντάλη, συντρόφισά μου, τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Αφιβάλλω λοιπόν και για τους στόχους τη κλιματική αλλαγή. Ε, βασική ερώτηση τώρα για την παραγωγή για ίδια κατανάλωση. Την πρώτη φορά που έγινε αυτό, εμεί, οι σοσιαλιστές εργαστήκαμε πάρα πολύ για να υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικέ που να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή ένδυα να κάνει προτάσεις και δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε όμως να είναι πιο φιλόδοξη η προσπάθειά σας κύριε Κανιέτε. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναπόκειται να το κάνει αυτό, όχι στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει οι στόχοι να είναι δεσμευτικοί και να έχουμε στόχους για την ενεργειακή απόδοση, υποχρεωτικούς και δεσμευτικού. Και κάτι άλλο που δεν αναφέρεται καθόλου είναι τα τέλη και οι φόροι. Ζητάτε διαφάνεια και εκεί. Αλλά δεν μπορεί να μετακυλείται όλο το κόστος στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού. Θα είναι ε, ε, απλησίαστη η ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες. Χαίρομαι για την πρόταση ε, για την παραγωγή προς ίδια κατανάλωση, αλλά η Ισπανική κυβέρνηση ακολουθεί άλλο δρόμο Κοιτάξτε, λέει η Πρόεδρο, κυρία Καπεθόν, όλοι θέλετε να κάνετε πολλέ ερωτήσει ε, και μετά πρέπει να απαντηθούν κι αυτέ. Αυτό είναι μια δυσκολία. Τι να κάνω κι εγώ. Είναι περίπλοκα τα πράγματα αυτά. Και οι ερωτήσει των συντονιστών ήταν περίπλοκε και απαιτούσαν μακροσκελεί απαντήσει. Όπω και αυτά που ρωτάτε εσεί τώρα. Την άλλη φορά θα ζητήσουμε από τον Επίτροπο να παραμένει περισσότερη ώρα μαζί μα, γιατί υπάρχουν τόσε πολλέ ερωτήσει. Ο κύριο Μπελέτ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με το είπε ο που απεχώρησε εδώ η εκδεξιόν Νομίζω ότι ήταν ε, ολοκληρωμένες εμπαντήσεις του Επιτρόπου και ε, απάντησε τόσες ερωτήσεις που δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε. Οπότε έχω απλώς μια γενική παρατήρηση. Έγινε πολλή κουβέντα όσον αφορά την φιλοδοξία της συμφωνίας στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και δεν συμφωνώ με την γενική άποψη, γιατί νομίζω ότι για το MSR έχουμε ξεχάσει κάτι. Το LRF. Και εδώ είχαμε τσακωθεί όσον αφορά αυτό το linear reduction factor. Και εσείς ε, συναδέλφισαν με τους συναδέλφους σας πώς ξεχάσαμε όλο αυτό το καυγά που κάναμε εδώ Θέλαμε να έχουμε πιο φιλόδοξη πρόταση από το Συμβούλιο για την ε, ε, αεροπλοή μεταφορές Άρα δεν ισχύει αυτό το βίβλο σαν γενική εντύπωση. Τώρα κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Εκτός μικροφώνου, λέει καλή κύριο Σέκφαρ. μπά, μπα. εσύ θα έπρεπε να είσαι στον για τι εκλογές. Μην κάνει εδώ εκλογέ. εκλογές. Εκλογές έχετε στο Άμστερνταμ, όχι εδώ. Να μην μεταφέρετε εδώ στο Στρασβούργο την πλοκή σας εκστρατεία. Και αυτό το 5% που αποτελεί βάση τη δική μας πρόταση που την έχει στηρίξει ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι εσύ δεν ε, ενέκρινε την πρόταση για το 5% αλλά όλες οι πτέρυγες ECR, ε, ΕΛΚ, σοσιαλιστές στήριξαν την πρόταση αυτή του 5%. Ίσως δεν το 5%, να μείνουν στο 2%. Ίσως στο μέλλον θα χρειαστεί το 5%. Ο μηχανισμός Duncan είναι στόχος για μη χρήση της ενέργειας. Ε, αυτό είναι φιλόδοξο, το υποστηρίξουμε, αλλά ίσω το Συμβούλιο δεν περάσει και μείνουμε στο 2%. Εσείς τι λέτε, θα περάσει το 5%? Ο κύριο Ντάμπλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλα τα ρωτήσαμε. Α, εγώ έλαβα το λόγο τελευταίο. Τέλο πάντων, κάτι άλλο θα ρωτήσω. Το ETS έχει εντοπίσει και το πρόβλημα. Πώ θα δούμε το ότι πολλέ φορέ μια πολιτική συγκρούεται με μια άλλη. Άρα να δούμε με ποιον τρόπο θα υπάρξει συνέργεια των πολιτικών και όχι σύγκρουση τους. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με τους σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Δώσατε την άδεια για ένα εργοστάσιο για πυρηνικά απόβλητα. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα με τον ποταμό Τάγο. Τι θα γίνει, πώς παίρνετε τέτοιου αποφάσεις. Χωρί να κάνετε διαπραγματεύσει με τι όμορε χώρε. Γιατί αυτό ο σταθμό που δώσατε απόφαση ήταν κοντά στα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πώ τι παίρνετε χωρί να υπάρχει. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ήδη εγώ έχω απαντήσει στην Επιτροπή και δεν πήρα απάντηση. Δεν ξεσήκωσα τον κόσμο, αλλά θέλω να μου απαντήσετε σήμερα, κύριε Επιτροπέ γιατί αυτό και του ε, Ευρωπαίου πολίτε, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν απαντήσει για τόσο σημαντικά θέματα. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Κέσσιγκερ. Mr. Faria. Α, όχι, κύριο Φαρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, ε, θα ήθελα να σας ε, μιλήσω σε σχέση με κάτι που είπε ο συνάδελφός μου για την ε, αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων. Αυτό είναι επονίδιστο. Ε, ε, η Ισπανική κυβέρνηση δεν ήρθε σε συνεννόηση με την Πορτογαλική κυβέρνηση, δεν έκανε τις περιβαλλοντικές μελέτες που όφιλε, δεν σεβάστηκε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ούτε τη Διεθνή. Εγώ ανησυχώ και για άλλα πράγματα. Παράδειγμα, ε, για την κατάσταση εξόριξης ουρανίου στην περιοχή της Σαλαμάνκα. οι ε, ε, παλιές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Μπούργος και στην Κορούνια. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά, κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε για τις εκλογές και εμείς θα έχουμε εκλογές στην Πορτογαλία και θα ήθελα να σας πω ότι... Ε, θέλω να σας συγχαρώ ασκήσατε πιέσεις στην αεροπλοεία για να υπάρξουν ρυθμίσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε πετύχει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, έχω μια ερώτηση και εγώ ετοιμάσει για τις αερομεταφορές, αλλά θα την αφήσω γιατί έχω καλυφθεί και να μιλήσω και εγώ για την πυρηνική ενέργεια και ιδιαίτερα να εκφράσω ανησυχίες σε πολίτες που διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές. Εάν παρατείνεται τη διάρκεια ζωής πυρηνικών αντιδραστήρων και δεν συμμετείχαν στην διαβούλευση οι γειτονικές χώρες. Ε, αυτό ισχύει και στα πλαίσια της Συνθήκης Ευρατόμ και της Οδηγίας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και πάντα έχουμε προσφυγές στα δικαστήρια από όμορες χώρες. Ε, ε, δύο ερωτήσεις λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, προτίθεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν κοντά σε παλιές πυρηνικές εγκαταστάσεις και πώς προτίθεστε να προωθήσετε τη συμμετοχή των πολιτών ε, σε αυτό το θέμα συζητήσει που γίνονται για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων. Κύριε Σχόγκαρ. Ευχαριστώ μια σύντομη ερώτηση στη μητρική μου γλώσσα. Τι γίνεται με την τελική τιμή που καταβάλει ο καταναλωτής βάσει της εμπειρίας μας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωστοί κανόνες και σε επίπεδο αρχών, ειδικότερα για ανθρώπους ε, που ε, καταβάλουν αρκετά υψηλό ποσοστό του εισοδήματος του οικογενειακού για, ε, για την ενέργεια. Σε ποιο βαθμό λοιπόν θα αλλάξουν οι τιμές. Και τι γίνεται με την ενεργειακή ένδυα και την κατάσταση στην Ευρώπη, συνεπώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, στον κανονισμό Λουλουσεφ. Ε, υπάρχει το άρθρο 8 που ασχολείται με το μέθοδο υπολογισμού για την απομάκρυνση των εκπομπών άνθρακα και λέγεται το νέο επίπεδο αναφοράς για τα δάση θα καθοριστεί βάσει της συνέχισης προηγούμενων πρακτικών και της ε, έντασης ε, της διαχείρισης των δασών όπως τεκμηριώθηκε ε, στην περίοδο από το 1990 μέχρι το 2009 για τα εθνικά δάση και την κατηγορία τους. Από το 1990 μέχρι το 1998 ένα μεγάλο κομμάτι της Κροατίας ε, είχε καταληφθεί από σερβικές δυνάμεις. Και τότε ε, η Κροατία δεν μπορούσε να ε, ασχοληθεί με τα καταληφθέντα δάση. Ακόμη και μετά τον πόλεμο δεν τα καταφέραμε λόγω των συνεπειών ε, των ε, προβλήματα με τα διάφορα που είχαν καταστραφεί και τις υποδομές που είχαν καταστραφεί. Ο υπολογισμός λοιπόν τη ένταση τη μελλοντική διαχείριση των δασών από το 2021 μέχρι το 2030 βάσει στοιχείων και δυναμική και ένταση εργασιών διαχείριση από την περίοδο που ξεκινά το 1990 αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση της Κροατίας. Θα προτείνα κάποιες τροπολογίες ώστε να γίνει κάποια εξαίρεση για την Κροατία και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους βουλευτές να μας υποστηρίξουν. Θα ήθελα να πείτε κύριε Επιτροπέ, η Κομισιόν θα δεχτεί αυτές τις αιτιολογίες που μόλις ανέφερα για την εξαίρεση αυτή την οποία προτίθεμαι να ε, ζητήσω για την Κροατία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Ζητώ συγγνώμη ε, γιατί θα δώσω μικρές απαντήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Ε, θέλω να απαντήσω με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οπότε ξέχασα να απαντήσω στην κυρία Ρωμάνο για τα δάση. ναι, συγγνώμη. Σίγουρα η διαχείριση των δασών θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη των κλιματικών μας στόχων. Υπάρχει στη Συμφωνία του Παρισίων και θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο διατάξεων του Λουλούσιεφ να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των δασών. Αυτό για να απαντήσω την τελευταία ερώτηση της συναδελφού που έφυγε η Κομισιόν θα αναλύσει τις τροπολογίες Συναδελφοί, θα, θα εξετάσει τις ε, ε τροπολογίες και θα τις ε, μελετήσουμε. Ε, κύριε Λαβέα, πρώην Πρόεδρε, είπατε τα προβλήματα αυτών που κατέβαλαν μεγαλύτερες προσπάθειες στην αρχή, που πέτυχαν καλύτερους στόχους. Είναι οπότε και σε καλύτερη θέση για να επιτύχουν και τους στόχους του 2030. Αλλά καταλαβαίνω τι λέτε, διότι είναι σαφές ότι ο επιμερισμός προσπαθειών εάν κάποιες χώρες δεν υπήρξαν οικονομικά ε, αποδοτικές ε, βρισκόντας σε διαφορετική θέση. Οπότε είμαι σίγουρος ότι στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν είναι αδυνατόν. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σα ε, και τα όσα αναφέρατε. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις για τη μακροχρόνια λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων. Απλά να σας πω ότι όπως έχουμε δημοσίευσει στην έκθεσή μας πέρυσι, η μακροχρόνια λειτουργία είναι πρόβλημα διότι απαιτεί ε, επενδύσεις 45 και 55 δισεκατομμυρίων σε επενδύσεις ε, η Κομισιόν δεν έχει άμεση αρμοδιότητα για την αδειοδότηση. Αυτές είναι αποφάσεις των κρατών μελών αλλά οι επενδύσει πρέπει να εκνοποιούνται στην Κομισιόν, η οποία πρέπει να εκδώσει γνωμοδότηση. Ε, ακούσα μια ερώτηση. από τον κύριο Φάρια για την περίπτωση της Πορτογαλίας. Απάντησα όλες τις γραπτές ερωτήσεις, ε, δεν ήταν μια-δυο, ήταν πολλές, τις έχω απαντήσει όλες, αλλά υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ισπανίας και Πορτογαλίας για την επίλυση του ζητήματος θα λάβετε τις απαντήσεις. Τις έχω δει. Ε, έχω μιλήσει με πολλούς Πορτογάλους ε, για αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, το ζήτημα. Και τώρα γίνεται συζήτηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων που πάει καλά, αλλά ε, η άποψη της Κομισιόν είναι πολύ σημαντική. Απαντήστε την ερώτηση, γιατί εμεί είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κόσμο θέλει να ξέρει Ε, ε, πρόκειται να λάβετε σύντομα την απάντηση. Την έχω δει. Μου τέθηκε μια ερώτηση για τα ηλεκτρικό, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι σαφές. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε ε, μόνο με την ε, ορισμό στόχων τη των εκπομπών. Χρειάζεται να βοηθήσουμε και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι ολιστική προσέγγιση μας. Στόχοι θα υπάρχουν. Θα είναι φιλόδοξοι Θα υπάρχουν σίγουρα στόχοι, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε πώς θα προωθήσουμε τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Ε, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων εντός των προτάσεων. Στο παρελθόν δεν λαμβάναμε υπόψη τα ηλεκτρονικά οχήματα καθόλου ε, για τη μείωση των εκπομπών ανθρακά. Στο μέλλον θα τα λαμβάνουμε υπόψη. Θα λάβουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους αυτή η πρόταση θα είναι πιο φιλόδοξη, πιο ολιστική και πιο ολοκληρωμένη και θα... Πριν τα τέλη του χρόνου, όσον αφορά τα ελαφρά και τα βαρέα οχήματα και τα αυτοκίνητα, ε, αυτά θα δούμε το 2018. Θα υπάρχουν διάφοροι στόχοι για τα οχήματα. Ε, μετά τις εκλογές. Όλα γίνονται πριν από, μετά από εκλογές. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για την εκτίμηση δικτύπου, διότι είναι περίπλοκη, πρέπει να αξιολογηθούν πολλά επίπεδα, πολλές ημερομηνίε, πολλά ορόσημα. Τι κάνουμε με τις παραμέτρους χρησιμότητας, το αποτύπωμα, πολλά στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη. εισαγωγή διαφορών στοιχείων και μου λέτε αν θα επιλέξουμε την πραγματική οδήγηση. Εμείς ζητάμε από όλους τους εμπειρογνώμονές μας να μας πούν πώς μπορούμε να κάνουμε ε, δοκιμές οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Δεν θα είναι σε αυτή την πρόταση, αλλά θα ανοίξουμε μια πόρτα για να εξεταστούν οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης, όπως έχουμε πει. Το μελετάμε. Υπάρχει το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Έχετε δει τα ολοκληρωμένα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Η φτώχεια είναι κομμάτι αυτού. Θα πρέπει να υποβάλλετε έκθεση ε, κάθε δύο έτη για την κατάσταση. Λαμβάνεται σε όλα τα σχέδια ενέργειας και κλίματος η ενεργειακή φτώχεια, σε όλους τους στόχους. Ζητάτε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ορισμό είναι περίπλοκο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα παρατηρητήριο που έχει ξεκινήσει τις εργασίες του αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί και πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με το κράτος μέλος. Είναι αρκετά περίπλοκο ορισμός, να υπάρξει ένας ενίος ορισμός για την ενεργειακή φτώχεια. Αλλά θα δούμε τις βελτιστές πρακτικές, τι έχει γίνει και θα... Κατά τη συζήτηση με τα κράτα μέλη θα δούμε ε, πώς προσεγγίζουν την ενεργειακή φτώχεια κατά κράτος μέλος. Επίσης είχαμε μια ερώτηση, μια πολύ περίπλοκη ερώτηση από την, την κυρία δεν ξέρω αν είναι εδώ, αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Ε, θα, τη γράψω, θα της γράψω γιατί χρειάζεται χρόνο. Με επέκρινε αρκετά και ο κ. Δούπεν ε, ε, κοιτά το ερώτημά του. Για τη συνοχή, ξέρετε, προσπαθούμε. Όταν κάνουμε την εκτίμηση προσπαθούμε κάθε μέτρο να έχει συνοχή με τα υπόλοιπα. Αρχικά. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, όταν πήγα να εξηγήσω το πακέτο, ε, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, ξέρετε γίνεται σε συνδυασμό με τα άλλα. Το πρόβλημα είναι ότι μόλις αρχίσει κανείς ε, να τροποποιεί τα πράγματα, χάνεται η συνοχή. Είναι περίπλοκο το εγχείρημα ε, και είναι δύσκολο εντό τη Επιτροπή. Ε, ξέρετε, έχετε το ETS, το ETS για την αεροπλοεία, την επιμερισμό ε, προσπαθειών και όλα αυτά, πώς αυτά συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση, την, τα ηλεκτρικά οχήματα. Αφού θα έχουμε ολοκληρώσει το πακέτο τη δέσμη μέτρων, θα προσπαθήσουμε, θα έχουμε κάποια συνοχή μέτρων. Ας ελπίσουμε ότι θα τη διατηρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ συνάδελφοι ε, που ήρθατε. Ε, κυρία Πρόεδρε, ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια παράκληση προς τον κύριο Επίτροπο για, να μου απαντήσει, γιατί δεν μου απάντησε θα το κοιτάξει ο Πίτροπο, θα το δείτε διμερώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη κύριε Πίτροπη, ούτε σε μένα απαντήσετε. Παρακαλώ να μου απαντήσετε για το θέμα των πυρηνικών αποπλήτων. Ναι, ε, λήξη συνεδρίαση. Ε, θα το δείτε διμερό, γραπτό κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.